Συνάδελφοι, δύο σύντομε ανακοινώσει. Πρώτα πρώτα θα πρέπει όλοι ε, να συμφωνήσουμε με αυτά τα οποία έγιναν ε, χθε και αυτά που είπε ο πρόεδρο Σούτς